Uh, Καλημέρα σας. Έχουμε αργήσει λιγάκι, καλό θα ήταν λοιπόν να ξεκινήσουμε. Με το σημείο 15 της μερίσας διάταξης, καθευθυντήριας γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2001, τμήμα 3. Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης ε, είναι μια καθοδήγηση για τον προϋπολογισμό του 2021. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο εισηγητής για αυτό το θέμα. Καλώς ήρθατε. Είναι το πρώτο στάδιο στην ε, διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2021. Το ψήφισμα και οι κατευθυντήριες γραμμές στην ουσία ε, δείχνουν ε, τις θέσεις του Κοινοβουλίου για τον επόμενο προϋπολογισμό που θα καταθέσει η Επιτροπή των Ιούνιων. Ε, η Επιτροπή του Προϋπολογισμού αποφάσισε να αλλάξει η διαδικασία του προϋπολογισμού εντός του Κοινοβουλίου και τώρα η κάθε Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να δίνει πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι που την αφορά κάθε φορά. Επίσης, η επιστολή για τον τριμερή διάλογο που ήταν η πρώτη αντίδραση της ΑΦΕΤ ε, μετά την ε, ανακοίνωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έχει επίσης αλλάξει. Ε, το 2021 είναι ένα ειδικό έτος σε επίπεδο προϋπολογισμού γιατί είναι και το πρώτο έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Υπάρχουν επίσης ε, μία σειρά νέων χρηματοδοτικών μέσων που θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στις αρχές του επόμενου έτους. Υπάρχει το μέσο για την ε, γειτονία και για την διεθνή συνεργασία και το ICI καθώς και το μέσο για την προενταξιακή βοήθεια. Οι διαπραγματεύσεις βέβαια και για τα δύο αυτά μέσα συνεχίζονται και μπορεί να επεκταθούν μέχρι και το δεύτερο ήμιση του έτους. Ε, ελπίζουμε ότι στις αρχές του επόμενου έτους ε, αυτά τα μέσα θα είναι διαθέσιμα και θα λειτουργούν. Ελπίζουμε όμως, περιμένουμε ακόμα ε, τις απαντήσεις σχετικά με το ΠΔΠ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα θα συναντηθεί προσπαθώντας να συμφωνήσει για το θέμα του ΠΔΠ. Αύριο το πρωί ε, ε, θα μάθουμε εάν έχει επιτύχει η προσπάθεια αυτή των ηγετών. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμφωνία ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο δεν πει το συντομότερο δυνατόν. Διότι αν Α στοχίσουμε σε αυτό, θα έχουμε καθυστερήσει στην εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών μέσων και γι' αυτό το Κοινοβούλιο επανειλημμένα ζήτησε από την Κομισιό να, ετοιμάσει σχέδια έκτακτη ανάγκη ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει χρηματοδοτικό κενό στι αρχέ του επόμενου έτου. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον εισηγητή για να παρουσιάσει το σχέδιο της γνωμοδότησής του. Κύριε Νίκο Ανδρουλάκη, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρουσιάζω σήμερα την νομοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021. Είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να εκφράσουμε τη γνώμη μας σε αυτό το αρχικό στάδιο και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μιλήσουμε για τις προτεραιότητές μας. Το 2021 θα είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου αλλά και της νέας αρχιτεκτονικής των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης. Για αυτό τον λόγο, στον περιορισμένο χώρο που είχα κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου που έχουμε, επέλεξα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχουμε από τα πρώτα στάδια προγραμματισμού και να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή για κάθε τρίτη χώρα που λαμβάνει σημαντικά ποσά στήριξης. Έτσι ώστε η δομή να μας επιτρέπει να εκπληρώνουμε αποτελεσματικά τον εποπτικό μας ρόλο. Καθώς σήμερα ξεκινάει η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι πρέπον να σημειώσουμε ότι χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και να πετύχει το στόχο της στρατηγικής αυτονομίας. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε περιοχές όπως είναι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και οι χώρες Ανατολικής Κοινότητας δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάμε τη σημασία που έχει η πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη χρηματοδοτική στήριξη. Επίσης, λόγω των περιορισμού λέξεων, θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες για ζητήματα τα οποία δεν μπορούσα να περιλάβω στο σχέδιο. Μεταξύ άλλων, σχετικά με το τρίτο μέσο για την προενταξιακή βοήθεια, το ύψος χρηματοδοτήσεων που θα λαμβάνουν οι υποένταξη χώρες θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των βασικών αρχών της Ένωσης, όπως είναι το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και οι σχέσεις καλής γειτονίας. Για τον λόγο αυτό και ιδιαίτερα όσο αφορά την Τουρκία, προτείνω τη μεταφορά όλων των διαθέσιμων κονδυλίων προ οργανώσει και ομάδε που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δράσει που επιτρέπουν τον απευθεία διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και προωθούν τι ευρωπαϊκέ αξίε. Τέλο, κάνω μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για την ανάπτυξη τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια, ζητώντα τον καλύτερο συντονισμό του και την ενίσχυσή του, ώστε να μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Η προθεσμία για τροπολογίε είναι αύριο στι 11 η ώρα. Περιμένω τα σχόλια και τι παρατηρήσει σα και είμαι σίγουρο ότι μαζί με του συναδέλφου θα μπορέσουμε να δημορφώσουμε μια πολύ καλή πρόταση προ την Επιτροπή Προπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα ήρθε η ώρα για τους σκιώδεις ε, να μιλήσουν. Ο κύριος Γκάλερ έχει ζητήσει το λόγο πρώτος. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, μας δίνει μια γενικότερη βάση, πολύ καλή βάση και συνάδει με τις ε, βασικές ιδέες μου. Επειδή έχω ασχοληθεί με την ασφάλεια και την ε, άμυνα τα τελευταία δέκα χρόνια και το έχετε τονίσει στην έκθεσή σας. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες τεχνικές και γεωγραφικές παρατηρήσεις και προσθήκες, για παράδειγμα. Πρέπει να τονίσουμε τη στρατηγική σημασία, όπως είπατε, της άμεσης γειτονίας των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής ε, ε, Ευρώπης ε, και της νότιας γειτονίας. Για άλλη μια φορά με αυτή την γνωμοδότηση μπορούμε να θυμίσουμε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι πρέπει να συνοδεύονται τα λόγια από πράξεις και να δίνονται τα χρήματα εκεί που πρέπει και να έχουμε συγκεκριμένες δράσεις στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυτές τις ημέρες ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συναντιέται, αύριο συγκεκριμένα θα έχει συνάντηση το Συμβούλιο για το νέο πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Ε, αν η Επιτροπή Φοντερ Λάιεν τον όλων των πολιτών δράσει ως σοβαρή γεωπολιτική Επιτροπή και μάθει όχι μόνο, και μάθει, όχι μόνο να μιλάει τη γλώσσα της γεωπολιτικής, ε, θα πρέπει το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε ως σχέδιο στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Η πρόταση του Σαρλ Μισελ βγάζει από τα ευρωπαϊκά project και ταΐζει τα εθνικά συμφέροντα. Ένα τέτοιο ΠΔΠ θα απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα υπερασπιστούμε τον κοινό μας ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τις επενδύσεις στο κοινό μας μέλλον, μακριά από εθνικούς εγωισμούς. Ε, πρέπει οι φιλοδοξίες να συνοδεύονται από δράσεις και οι δράσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται σωστά. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτή τη γνωμοδότηση ε, θα μπορέσουμε ε, τα σημεία αυτά των απόψεών μας να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο σκιώδη. Οπότε είναι η σειρά των ε, ευρωβουλευτών να μιλήσουν. Ο κύριος Μπασέσκου έχει το λόγο. Παρακαλώ. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά σχόλια. Μόνο μία παρατήρηση. Proposal, του... Σχετικά με την Τουρκία. Η πρόταση να ακυρωθούν ε, τα κονδύλια για την Τουρκία δεν είναι, θεωρώ, η καλύτερη ιδέα. Δεν θα δώσω κάποια εξήγηση ε, και ούτε θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Τουρκίας. Απλώς ε, λίγα λόγια να πω. Όλοι μας κατηγορούμε την Τουρκία για την ε, επέλασή της ε, στη βόρεια Ανατολική Συρία. Πιθανόν γι' αυτό ο συνάδελφος ε, προτείνει να ακυρωθεί η χρηματοδότηση για την Τουρκία. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία Ε, το να απομονώνουμε τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία ε, ε, ε των του Κούρδων, εντάξει αυτό θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν υποστηρίζω βέβαια αυτή την ιδέα, όμως ε, είναι μια παρέμβαση που κάνει και είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας. Θέλει να απομονώσει τη χώρα από της τις ροές των Κούρδων. Αυτό ε, βέβαια ο εισηγητής τι να έχει πιο ισχυρή γνώμη, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Το να απομονώσουμε την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι λάθος. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον που να θέλει το λόγο. Επομένως, επανέρχομαι στον κύριο Ανδρουλάκη για τη δευτερολογία του και για να απαντήσει στις ε, απόψεις που ακούστηκαν τώρα. Δεν είναι μόνο ε, η εξωτερική πολιτική. Προφανέστατα τα όσα συμβαίνουν στη Συρία έχουν ε, όλους μας προβληματίσει πάρα πολύ, διότι είναι ένας πολύ σκληρός εμφύλιος με εκατομμύρια πρόσφυγες και θέλαμε όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται να είχαν μια άλλη στάση για τα πράγματα. Είναι πάνω απ' όλα όμως τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το κράτος δικαίου, και χαρακτηριστικό παράδειγμα ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τι προηγούμενε μέρε τι έγινε τον κύριο Καβάλα, όπου λίγε λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή του ξανασυλλήφθη ω τρομοκράτη με την αδίθεν εμπλοκή του στο πραξικόπημα. Άρα δεν έχει να κάνει τόσο όσο με το θέμα της Συρίας, έχει να κάνει με το εσωτερικό και με τις ευρωπαϊκές αξίες. Άποψή μου είναι, και πιστεύω είναι και άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι οι χώρες που έχουν φάκελο πρόοδου, που ένταξη χώρες, πρέπει να σέβονται το βασικό πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών. Thank you, Ευχαριστώ. Ο κύριος Πασέσκου θέλει να επανελθεί. Όχι. Ναι. Ε, πρόεδρε, απλώς να χαιρετήσω την άποψη του εισηγητή χωρίς να αλλάζω τη δική μου. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι αύριο στις 11. Κλείνουμε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο. Το σχέδιο σύστασης για τα Δυτικά Βαλκάνια εν ώψη και τη συνόδου του Ζάγκρεμπ για το Μάιο φέτος. Αυτή η έκθεση έρχεται στο πλαίσιο της ε, επανεξέτασης της ε, μεθοδολογίας για τη διεύρυνση για Αλβανία και Βόρειο Μακεδονία και το σχέδιο επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια όπως και τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται εν εξελίξη για την προενταξιακή βοήθεια και η οποία θα κατευθύνει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή στην περίοδο 21-27. Ο κύριος Πιτσούλα έχει το λόγο, ο εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Πολύ με ευχαριστεί αυτή η δυνατότητα να σας παρουσιάσω το σχέδιο συστάσεων εν ώψη της συνόδου όπως είπατε κι εσείς. Ήθελα να τονίσω ότι η βασική πρόθεση με την έκθεση αυτή ήταν να στείλουμε καθαρά πολιτικά μηνύματα ώστε να επανενεργοποιήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης και τη συνέχεια της. Άλλο βασικό μήνυμα είναι η μεταρρύθμιση της Ένωσης που θα πρέπει να τρέχει παραλλήλως προς τη διεύρυνση η εσωτερική πολιτική κατάσταση στα κράτη-μέλη δεν μπορεί να είναι λόγος διακοπής ή αναστολής της διαδικασίας. Μιλούμε για μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ένωσης από την αρχή, από την δημιουργία της, ώστε να επεκτείνεται η περιοχή της δημοκρατίας, της ευημερία και της ειρήνης. Επενδύσεις στην αμοιβαία ασφάλεια και ευημερία έχουν ε, σίγουρα συνεισφέρει προς την ε, ειρήνη σε πολύ μεγάλες εδαφικές περιοχές. Πρέπει να σκεπτούμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Η λανθασμένη κατά την άποψή μου άποψη να μην ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, ε, έχει αντίκτυπο και συζητείται στις πρωτεύουσε εμείς ζητούμε να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες αυτές ήδη το Μάρτιο. Η νέα πρόεδρος και ο ύπατος εκπρόσωπος έχουν δηλώσει ότι η νέα επιτροπή στοχεύει στην γεωπολιτική της παρουσία. Πρέπει αυτό να το αποδείξουν με πράξεις και ο πιο εύκολος τρόπος θα ήταν στην άμεση γειτονία μας. Το σχέδιο υποστηρίζει ε, τις ιδέες που επεξεργάστηκαν οι Επιτροπές ε, Επικοινωνίας για διαβριμένη μεθοδολογία, ανοιχτά κεφάλαια και δέσμες, εξασφαλίζοντας τις περιοχές πολιτικής και τις ε, ποιοτικέ μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα, ώστε να έχουμε αυτά αποτελέσματα στις χώρες διαβρύνσης, επιτρέποντας παράλληλες διαπραγματεύσεις σε διάφορα κεφάλαια και πιο συνεπή κριτήρια αξιολόγησης και συνεχιζόμενη υποστήριξη σε όλη την διαδικασία, όπως και καταμέτρηση, εξακρίβωση δηλαδή της πρόοδου, ώστε να αξιολογείται κάθε χώρα επί τη βάση των δικών της ικανοτήτων. Η υλοποίηση της διαβημένης μεθοδολογίας για τις χώρες διεύρυνσης θα πρέπει να διευκολυνθεί. Μόνον εφόσον βεβαίως οι χώρες αποφασίσουν να έχουν να συμμετάσχουν. Το να αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο στον τίτλο της ανακοίνωσης δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Το Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί να υποστηρίξει τις δημοκρατικές διαδικασίες στην περιοχή και να βοηθήσει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην ενταξιακή τους πορεία. Έχουμε συζητήσεις και επαφές με κάθε χώρα διεύρυνσης εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες και μπορούμε να συνεισφέρουμε στις προσπάθειες αυτές και επομένως εισάγουμε και κάποιες από τις νέες προτάσεις όπως την ειδική πλειοψηφία σε ανοιχτά και κλειστά κεφάλαια και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία αναστολής. Ε, περιμένουμε το Ζάγκρεμπ, Σύνοδος, να επιφέρει πρόοδο για την ε, συζήτηση και την οικονομική πρόοδο να υπάρξει συμφωνία υποστήριξης της διαδικασίας διεύρυνση για το μέλλον. Τέλος, το σχέδιο έκθεση έχει και έναν περιορισμένο χώρο των συστάσεων. Θα υποβάλω και εγώ ίδιο τροπολογίες για να επεκτείνω το περιεχόμενο και εδώ βασίζομαι στην ε, επικοδομητική συνεισφορά των ε, σκιωδών και των ε, συνεισηγητών. Ε, υπάρχει κάποιος άλλος ε, που ζητάει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Πιτσούλα για, την, ε, για το σχέδιο. Νομίζω ότι όλα αυτά που χρειάζονταν υπάρχουν στο κείμενο και συμφωνώ και εγώ με την αποστολή σαφούς μηνύματος και συστάσεων είναι καλό να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για τα Δυτικά Βαλκάνια, διότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται. Εγώ συμφωνώ απολύτως με κάποιες παραγράφους του κειμένου που ίσως να μην είναι στην ε, κεντρική συζήτηση που διεξάγεται σήμερα, τη σημασία περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες, στις υποδομές, στην ανάπτυξη κτλ. Βεβαίως και θα υπάρξουν τροπολογίες από πλευράς μου και από πλευράς των συναδέλφων, αλλά με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω την έκθεση, αναλόγως προς τα όσα ανέφερε και ο κύριος Πιτσούλα. Η ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να αναφέρεται ως τέτοια στις συστάσεις, αλλά έχω δύο ερωτήσεις που δεν μου ήταν απολύτως σαφής. Σαφή τα στοιχεία αυτά δηλαδή στην έκθεση. Τι εννοείται στο σημείο α ότι η εσωτερική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διεύρυνσή της λέτε and its enlargement ότι αυτά πρέπει να τρέξουν παραλλήλως και στο F ότι η καλύτερη συνέπεια μεταξύ της διεύρυνσης και των πολιτικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πώς μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει, τι εννοείται με αυτό. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή. Ο κύριος Κιούτσου από τους Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πίτσουλα, για την εξαιρετική προετοιμασία αυτής της πολύ θετικής σύστασης, θα έλεγα σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια ε, και την ε, Σύνοδο Κορυφή ε, του 2020. Είναι καλό που έχουμε τελικά μια απτή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με μια νέα μεθοδολογία η οποία θα αφαιρέσει τις ανησυχίες των χωρών που αντιτίθεντο σε αυτή την διεύρυνση και θα δώσουμε έτσι μια νέα όθηση στην διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ήδη μια περίπλοκη διαδικασία. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά τις ευρωπαϊκές προσδοκίες ε, των λαών των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, αυτά φαίνονται στο κείμενο και γι' αυτό ε, να πω ξανά ότι ε, υποστηρίζω την άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, άλλος, καθώς και τη συζήτηση με το Κωσυφοπέδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή του προοπτική. Η ομάδα μου έχει ε, μια πολιτική για τα Δυτικά Βαλκάνια την οποία ε, βασίζει στην κατανόηση. Αυτό φαίνεται στην έκθεση του κυρίου Πίτσουλα. Αυτά πρέπει να γίνονται σε συνδυασμό με τη διαδικασία διεύρυνσης. Ευχαριστούμε. Το ECR και η κυρία Φωτέγκα έχουν το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πίτσελα για την ε, πολύ καλή αυτή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ για τις διαπραγματεύσεις ε, με τους σκιώδεις ε, και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτές. Παρόλο που έχω διαφορετική άποψη για κάποια από τα θέματα, Σίγουρα βλέπω το θετικό, πολύ θετικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνουμε γενικότερα. Υπήρξε μία περίοδος απεσιοδοξίας μετά την έναρξη της προηγούμενης νομοθετικής περίοδου και ειδικά ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες περιοχές Είχαμε πολύ άσχημα σήματα που, και μηνύματα που στείλαμε στους εταίρους μας. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους φραγμούς ε, που υψώθηκαν στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και ελπίζω ε, η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει με επικοδομητικές προτάσεις ε, που θα επιδιώξουν την διεύρυνση. Ειδικά για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, να πω ότι έχουν και οι δύο χώρες καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ε, για να εκπληρώσουν τα, τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ο ηγέτης της Βόρειας Μακεδονίας ε, ε, μπήκε σε πολλούς πολιτικούς κινδύνους προκειμένου να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τον στηρίξουμε. Να τονίσω ότι ε, για τη δική μας ομάδα το ε, και είναι ένα, μια κόκκινη γραμμή και θα ήταν λίγο επικίνδυνο να το βάλουμε αυτό μπροστά. Ευχαριστώ. Κύριο Κιούτσεκ θέλει να προσθέσει κάτι. Ε, ένα τεχνικό αλλά πολιτικό ε, σημαντικό θέμα. Είχαμε μια συμφωνία με τον εισηγητή. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες μέρες μέχρι τις τροπολογίες. Μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την προθεσμία μέχρι τις 2 Μαρτίου, διότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι πράσινη εβδομάδα, θα βρίσκονται αλλού οι συνάδελφοι. Νομίζω είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε ένα στιβαρό κείμενο στη διάθεσή μας. Δελαβαίνουμε ότι ο κύριος Πιτσούλα το δέχεται. Μέχρι πότε είπατε, 2 Μαρτίου. 2 Μαρτίου τότε. Στις 11 η ώρα πάλι. Ε, Basescu like to speak. Ο κύριος Μπασέσκου θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω μερικά σχόλια. Πρώτον, σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης που γνωρίζουμε όλοι έχει επιταχυνθεί κατά τη περίοδο των διαπραγματεύσεων. Ένας ε, στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση της οικονομίας για να επιτευχθεί ε, το λεγόμενη ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς. Πιστεύω, με βάση την εμπειρία μας, είτε μιλάμε για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Τσεχία, η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να γίνει αφού, αφότου οι χώρες έχουν ε, γερά ε, δικαστικά συστήματα ε, γιατί θα, η διαφθορά κατά διάρκεια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης θα είναι πραγματικότητα και μετά θα τους ζητάμε να καταπολεμήσουν τη διαφθορά αλλά εμείς τους οθούμε πρόημα να ιδιωτικοποιήσουν τις οικονομίες τους πράγμα που Συνέβηκε τουλάχιστον στη Ρουμανία. Δεν θα μιλήσω για άλλες χώρες. Δεύτερη παρατήρηση. Σχετικά με τους πρόσφυγες. Τους κάνουμε μια εξαιρετική σύσταση να συνεργαστούν με τη Frontex, με τον Frontex. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την άποψή μου, οποιαδήποτε συνεργασία με τον Frontex θα έχει λιγότερα αποτελέσματα από ό,τι εμείς αναμένουμε εδώ. που μιλάμε εδώ με θεωρητικούς όρους, στην πράξη θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, ε, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα στα ε, κυκλώματα της μετανάστευσης. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τις συμφωνίες επανεισδοχής, να την ε, οριστικοποιήσουμε αυτές με τις χώρες που διοχετεύουν μετανάστευση, με τις χώρες διαμετακόμισης, συνεργασία με τις κυβερνήσεις έτσι ώστε να εξουδετερώσουμε το οργανωμένο έγκλημα που ε, δημιουργεί αυτό αυτές τις μετακινήσεις και τέλος να αναχαιτήσουμε ε, τα πλοία που μεταφέρουν τους μετανάστευση. Τώρα τους δίνουμε σύσταση να συνεργαστούν με το Frontex. Αυτή η σύσταση δεν είναι σοβαρή προσέγγιση διότι έχουμε την εμπειρία. Ο Frontex δεν μπορεί να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση. Και τέλος, σχετικά με τη διαρροή ε, εγκεφάλων, τη διαφυγή εγκεφάλων. Τι να κάνουμε για αυτό το θέμα. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή. Η Ρουμανία έχασε 16.000 γιατρούς και 220.000 μηχανολόγους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τι, τι, τι συστάσεις κάνουμε τώρα σε αυτές τις χώρες. Okay. These were my uh, observations. Αυτές τις παρατηρήσεις είχα. Πιθανότατα να προτείνω κάποιες τροπολογίες προσπαθώντας να βρω κάποιες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Βλέπω έναν άλλο σκιώδη από τους περάσινους, η κυρία Βιόλα Φων Κράμον, το Μπάτελ. Θα θέλατε να ε, σχολιάσετε την έκθεση Πιτσούλα. No. Thank you, Chair, uh, for Ευχαριστώ που μου δίνετε στο καθυστερημένο αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή την έκθεση. Ε, ε, είδα ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη προσδοκία για τη διάσκεψη επέστρεψα από το Βιλγάρι χθε το βράδυ και όλοι μιλάνε για τη τελευταία διάσκεψη κορυφή και την υποχρέωση του Ευρωκοινοβουλίου να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι σίγουρο. Κάτι άλλο. Νομίζω όλοι συμφωνούμε με τις επικείμενες πιέσεις, ιδιαίτερα από τις κινέζικες επενδύσεις στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα στη Σερβία αυτό είναι πρόδειλο, είναι εμφανέστατο. Υπάρχουν μεγάλοι, μεγάλες εταιρείες, μεγάλες παίκτες εκεί ε, στον τομέα της οικονομίας. Αυτό μας δυσκολεύει την κατάσταση, ενώ εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε τις ίδιες συνθήκες που προσφέρουν κάποιες κινέζικες εταιρείες ή και το κινέζικο κράτος. Αυτό έχει σημασία και απασχολεί πολλούς ανθρώπους όχι μόνο της αντιπολίτευσης ή το πιο επικριτικό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά και ε, στους κόλπους της κυβέρνησης. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρότερη ανταπόκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, ε, μια... Ε, ισχυρότερη ανταπόκριση. Η μεθοδολογία γενικώ ε, παρουσιάζεται με θετικό τρόπο, υπάρχει μεγάλη ελπίδα. Ωστόσο, ε, υπάρχει κάποια ασάφεια στο ποσό της, του επενδυτικού σχεδίου προς τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήταν καλό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, να έχουμε κάποιο φιλόδοξο νούμερο, γιατί αν θέλουμε να επιφέρουμε αλλαγές στην κλιματική αλλαγή, ε, στην εξάλληψη του άνθρακα, θα πρέπει ε, να έχουμε μια ελκυστική προσφορά σε αυτές τις περιφέρειες για το πώς να ε, υπερπηδήσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Εκεί περιμένουν και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας. Ε, βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Green Deal ήδη έχει, κάποια, ε, έχει θέσει κάποια ερωτηματικά. Εναπόκειται σε εμά να εξηγήσουμε τι ακριβώς θέλουμε, τι περιμένουμε και τι θα μπορούσαμε εμείς να προσφέρουμε σε ό,τι αφορά νέες επενδύσεις, νέες ε, τεχνολογικές έρευνες και ειδικά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης το η κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι πολύ άσχημη στα περισσότερα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, με τη μορφή επιχορηγήσεων κρατικών ε, σε ό,τι φορά την υγεία, το αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αν δεν επιλύσουμε ε, την ατμοσφαιρική ρήπανση. Ε, αυτό θα είναι ένα πολύ μακροπρόθεσμο πρόβλημα για όλη την περιφέρεια, αλλά και για άλλες χώρες όπως είναι η Σλοβενία, η Κροατία και η Ρουμανία, χώρες μέλη μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να, έχουμε κα... να είμαστε πιο φιλόδοξοι στο να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Στη σημείωσή μου έχω ε, ε, τον κύριο Άλαν Τζόνς από την DG Near. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα-δύο σχόλια και από μένα. Εμείς χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή, που είναι μια σαφής και ενθαρρυντική συνεισφορά σε πολύ κέριο χρονικό σημείο. Εμείς δουλεύουμε επί τριών αξώνων για τα θέματα διευρύνση. Καταρχά έχετε δει την ανακοίνωση για την ε, αναθεωρημένη μεθοδολογία της 5 η ε, Φεβρουαρίου για το άνοιγμα διαπραγματεύσεων με Αλβανία και Βόρειο Μακεδονία θα επανέλθουμε με επικαιροποιημένα σχόλια για να βοηθήσουμε τη συζήτηση αυτή και ως προς την σύνοδο του Ζάγκρεμ για την ε, οικονομική ανάπτυξη της ε, περιοχής, η αναθεωρημένη μεθοδολογία προσπαθεί να καταστήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική επί τη βάση της αξιοπιστίας, της προβλεψιμότητας και της ε, αυξημένης δυναμικότητας. Επίσης υπογραμμίζουμε τα ουσιαστικά στοιχεία των βασικών μεταρρυθμίσεων, των δημοκρατικών θεσμών, και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Πρώτη συνόδου ε, τέλη Μαρτίου κατά πάσα πιθανότητα θα επανέλθουμε με μια ανακοίνωση με ιδιαίτερη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επενδύσεις, καλύτερη συνδεσιμότητα και καλύτερη χρήση των ευκαιριών της ε, Πράσινης Συμφωνίας και του Πράσινου Θεματολογίου. Και στο σχέδιο έκθεσης ε, υπάρχουν πολύ χρήσιμες συνεισφορές προς την κατεύθυνση αυτή και ευχαριστούμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι η ΕΔ, η κυρία Φένετ, που είναι επικεφαλής ε, του Τμήματος Δυτικών Βαλκανίων, εκπροσωπείται. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς Είμαστε απολύτως υπέρ της ε, πρωτοβουλία του περιεχομένου του σχεδίου έκθεσης, όπως ε, είπε και ο συνάδελφος ε, της Επιτροπή, και εμείς συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της αναθεωρημένης μεθοδολογίας και συμφωνούμε στην γενική κατεύθυνση. Έχουμε δυόμιση μήνες τώρα για τα παραδοτέα αυτά, ώστε το Ζάγκρεπ να είναι επιτυχές, επιτυχία και νομίζω ότι πρέπει να εστιαζόμαστε διαρκώς και στις πολιτικές μας δεσμεύσεις ε, για τι ε, περιοχές, γιατί έχουμε δει και με τις συναντήσεις και επαφές που είχαμε και με όλους τους ομιλητές και με την άτυπη συνάντηση στο Συμβούλιο, ο ύπατο εκπρόσωπος, ε, η διάσκεψη του μονάχου για την ασφάλεια, όλα αυτά τα μηνύματα είναι πολύ σημαντικά στην προετοιμασία της Συνόδου του Ζάγκρεμ και θα χαιρέτιζα εδώ και το ρόλο του εισηγητή και των αντιπροσωπιών στις επαφές με τους ομολόγου μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό μήνυμα για το πώς συνεργαζόμαστε με τα Δυτικά Βαλκάνια στο ευρύτερο πολιτικό θεματολόγιο, κλιματική αλλαγή, πολυμέρεια, μετανάστευση, ε, πολιτική άμυνα και ασφάλεια, καλύτερη ευθυγράμμιση πρώτη διεύρυνση και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους ομολόγους μας στα Δυτικά Βαλκάνια ώστε να υπάρξει όλο και μεγαλύτερη προσέγγιση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής για τα θέματα μετανάστευσης. Είμαστε υπέρ της ολιστικής προσέγγισης, λέει η ομιλήτρια, επί ιδιώδων ροών και τα λοιπά, αλλά και άλλοι οργανισμοί και άλλες υπηρεσίες από την αρχή ας πούμε τις λειτουργίες της Frontex ε, στα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε δει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά θα είχα να προσθέσω στη συζήτηση, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθω στον κύριο Πίτσουλα. Ε, έχετε κάποιες απαντήσεις, κάποιες παρατηρήσεις ε, τελικές. Θα προσπαθήσω και τα δύο, Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω <clears throat> τους συναδέλφους για τις ε, παρατηρήσεις τους, ε, τις ερωτήσεις. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και θα τα λάβω υπόψη μου. Κάποια από αυτά βεβαίως ε, θα είναι αντικείμενο της περαιτέρω συζήτησης, λέει ο μιλτής. Για την ερώτηση της κυρίας Κίνγκ. Δεν θα έπρεπε να είναι δίλημα το θέμα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να ανανεώνεται, να μεταρρυθμίζεται και να διευρύνεται εξωτερικά. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προσαρμοστεί, να ανταποκριθεί προς τις προσδοκίες των πολιτών και γι' αυτό έχουμε και τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αναθέσαμε στον εαυτό μας να το κάνουμε αυτό, να το έχουμε κάνει μέσα σε μια διετία. Ποιος είναι ο στόχος της διάσκεψης για τα μέλλον της Ευρώπης. Ακριβώς να προσαρμόσουμε τους θεσμούς μας, να κάνουμε τα προγράμματά μας πιο αποτελεσματικά, να διευκρινίσουμε τις προθέσεις μας για την επόμενη εντολή να είναι όλα αυτά πολύ σαφή για τους πολίτες. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε και μάλιστα να τα κάνουμε καλά. Τώρα, παρά τα ενθαρρυντικά νέα από κάποια κράτη-μέλη, βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό που είχε αποκαλέσει ο πρόεδρος Γιούνκερ ζώνη ιστορικού λάθους. Περιμένουμε το Συμβούλιο του Μαρτίου να διορθώσει ή όχι το σφάλμα του Οκτωβρίου και πρέπει να περιορίσουμε και το περιθώριο στρατηγικών εκπλήξεων. Πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι, πρέπει να είμαστε υποστηρικτικοί της διαδικασίας διεύρυνσης που είναι ζωτική σημασία για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 21ο αιώνα και συμφωνώ απολύτως με εκείνους τους συναδέλφους που δικαίως μας λένε <clears throat> ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ αποτελεσματικούς ανταγωνιστές στα Δυτικά Βαλκάνια. <clears throat> Πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τις κεντρικές αξίες και αρχές μας. Πρέπει να επιδιώκουμε διαρκώς καλύτερη διακυβέρνηση, διοίκηση και να ενθαρρύνουμε τους εταίρου μα στα Δυτικά Βαλκάνια να αντιμετωπίζουν έτσι τάσεις μεγάλης κλίμακας και αρνητική ίσως σημασίας, δημογραφικέ τάσει, την αποτελεσματικότητα των θεσμών, το οργανωμένο έγκλημα, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, του οικοστήματος προσπαθούμε από αυτά τα ευρύτατα προβλήματα να συμπεριλάβουμε ό,τι μπορούμε στο κείμενό μας προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι πιο εμφανές στην διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον στην επόμενη συζήτηση των σκιωδών. Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά να σας θυμίσω ότι 2 Μαρτίου στις 11 η ώρα είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Τώρα θα κάνουμε για λίγα λεπτά ένα διάλειμμα για να περιμένουμε τον ειδικό εισηγητή Πέτρας Αουστρεβίτσιους, ε, ώστε να ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με το πρόγραμμα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 10 και 20. Επειδή όμως βλέπω πως όλοι είμαστε εδώ, ας ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η σύσταση προς το Συμφούλιο, την Επιτροπή και τον είπα το εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου του 2020 από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρονιά αυτή θα σηματοδοτηθεί από την Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο για την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει μια σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον κύριο Μπορέλ, πρόεδρο, είπα το εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επίσης, το Γενάρη είχαμε μία επικοδομητική ακρόαση. Αδειμονώ λοιπόν για την ανταλλαγή απόψεων και ξεκινώ με τον εισηγητή Πέτρας Αουστρεβίτσιους από το Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Να θέσω υπό την προσοχή σας την σύσταση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον είπα το εκπρόσωπο της Ένωσης ε, ε, για θέματα ανατολικής εταιρικής σχέσης εν της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου του 2020. Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε την πρωτοβουλία για την ανατολική εταιρική σχέση ε, μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις σχέσεις της με τις ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Καταρχάς γιατί η ανατολική εταιρική σχέση αποδείχτηκε ένα μέσο πολιτικής κινητοποίησης. Δεύτερον, λειτουργήσε ως μεγάλο κίνητρο για ολοκληρωμένες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και τρίτον, σηματοδότησε μια αλλαγή, μια στροφή ε, στα θέματα της ε, ε, ανατολικής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε τις αρχές για τη μελλοντική συνεργασία μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτραβήξει τη χείρα βοήθειας και συνεργασίας από τους, Ανατολ... τους γειτόνους μας στην Ανατολή. Οι βαθιές ολοκληρωμένες ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου βοήθησαν ε, να μπούμε σε ένα νέο στάδιο ε, σχέσεων με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία συγκεκριμένα. Η αυξημένη πολιτική συνεργασία και η εκτεταμένη οικονομική συνεργασία, οι εμπορικές σχέσεις έδωσαν τη δυνατότητα στις έξι ε, χώρες ε, της ανατολικής γειτονίας να γίνουν ο δέκατος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Μεγάλο επίτευγμα αν λάβετε υπόψη την ε, υποτονική οικονομία στις χώρες αυτές και τις προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι οικονομίες τους. Να συνοψίσω λέγοντας ότι οικονομικά όλο και περισσότερο αλληλοσυνδεόμαστε και αλληλοεξαρτόμαστε. Αυτή η μεταρρυθμιστική ισχύς ε, οδήγησε τις χώρες ε, της Ανατολικής Γειτονίας ε, σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εναρμόνιση και streamlining πολλών τομέων. Για παράδειγμα, στον τομέα του φυσικού αερίου. Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τη μεταρρύθμιση ε, του unbundling της αποσύνδεσης των διαφόρων τομέων. Η Ναυτογκάς έγινε, ε, είναι η μεγαλύτερη βέβαια εταιρεία στην Ουκρανία, όμως βγήκε από μια μεγάλη μαύρη τρύπα και έχει γίνει τώρα ο μεγαλύτερος ε, ε, φορολογούμενος της χώρας και δίνει μέρισμα σε όλους. Ε, έχουμε πολλές ιστορίες ε, ε, που είχαν ακουστεί για διαφθορά. Τώρα η ναύτογκας αποτελεί πολύ σημαντική επιτυχία σε οικονομικό επίπεδο. Οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας χρειάζονται μεγαλύτερη ενίσχυση ε, για να προχωρήσουν στην καινοτομία. Καταρχάς, η συνεργασία μας πρέπει να είναι υπό όρους. Να υπάρχει ε, πολιτική ελευθερία, κράτος δικαίου, ε, θεμελιώδη δικαιώματα και όχι διαφθορά. Δεν θα πρέπει αυτοί οι όροι και οι αρχές να θυσιαστούν μόνο και μόνο στο βωμό των οικονομικών κερδών. Δεύτερον, θα πρέπει η υποστήριξή μας για την ανοικοδόμηση του κράτους και των θεσμών ε, να γίνεται μέσα από ε, δράσεις ε, πολύ συγκεκριμένες και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες απειλές ασφαλείας και υβριδικές απειλές στις χώρες αυτές. Τρίτον, οι χώρες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο η καθεμία να υπάρχει περισσότερη ε, ευθύνη και ε, ιδιοκτησία ως προς την πολιτική ανατολικής γειτονίας από την πλευρά τους. Να είμαι λοιπόν αισιόδοξο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την αρχή less for less για αυτές τις χώρες, ε, λιγότερα για λιγότερα δηλαδή. Το more for more, το περισσότερα για περισσότερα θα είναι η βασική μας αρχή της επόμενες, στο επόμενο διάστημα. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη σύνταξη του πρώτου σχεδίου των συστάσεων μας έγινε μια συζήτηση για κάποια θέματα σε επίπεδο δομής, ε, ξεκάθαρα και καλά δομημένα τμήματα. Ε, το πρώτο έχει να κάνει με τον διαρθρωμένο διάλογο, την ενοικοδόμηση του κράτους ε, και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ζητούμε λοιπόν να γίνουν και άλλες προσπάθειες στην οικονομική συνεργασία και την νομοθετική εναρμόνιση. Προτείνουμε επίσης κάποιες καινοτομίες που θα έρθουν από τις ε, τροπολογίες ε, και από τη συζήτησή μας ε, για τη χρήση των νέων μέσων και την περαιτέρω επέκτασή τους. Για παράδειγμα, η αδελφοποίηση. Και φυσικά δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ολοκλήρηση της μεταρρύθμισης ε, του δικαστικού ε, σώματος ε, και της, και της διοίκησης. Στον τομέα της οικονομικής πολιτικής έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στην περαιτέρω ρυθμιστική σύγκληση σε πολλούς τομείς και για να είμαι ειλικρινής και ξεκάθαρος. Πιστεύω ακράδαντα στον κοινό οικονομικό χώρο με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Η εταιρική σχέση στον οικονομικό τομέα πρέπει να οδηγήσει σε ολοκλήρωση έτσι ώστε με τους όρους που έχουμε θέσει να έχουμε μία ανοιχτή αγορά με τους ε, εταίρους μας ε, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως ε, σε αυτό το τομέα. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται ως μεγάλη πρόκληση και μεγάλη απέτηση, όμως ε, αν γίνουν οι ολοκληρωμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις ε, ε, που προτείνουμε, οι χώρες αυτές θα μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή. Επίσης, η κεφαλαιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, η δημιουργία ανθρωπίνου κεφαλαίου, θα λαμβάνει υπόψη της σοβαρής κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές ε, λόγω της ε, μετανάστευσης του πληθυσμού τους, χάνουν πληθυσμό. Όμως θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό με μεγάλη μου χαρά βλέπω το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να ιδρύεται στην όμορφη πόλη του Κιέβου. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της συμμετοχής μας ε, ε, στον ακαδημαϊκό τομέα. Ε, εμείς φέρνουμε τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην Ουκρανία και τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Επίσης αυξάνουμε τη συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών γιατί τους θεσπίζουμε ένα κοινό πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Επίσης, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Να, ένας τομέας ε, στον οποίο θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Πέντε στους έξι ανησυχούν για την ασφάλεια και για τις σειράξεις. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να αντιμετωπίσουμε με το σωστό τρόπο, τρόπο τις ανησυχίες και τα θέματα που προκύπτουν εξαιτία αυτού. Θα πρέπει να εξετάσουμε ε, μια στρατηγική για την προπαγάνδα, το οργανωμένο έγκλημα, ε, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και κάθε είδους εγκληματική ενέργεια γενικότερα. Ποτέ δεν θα έρθει η βοήθεια ε, σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Και για τις επικοινωνίες, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για τις ε, επιτυχίες μας, τα επιτεύγματα που είχαμε στη συνεργασία μας με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Έγινε μια καλή αρχή, πολλά έπονται και πρέπει να επικοινωνήσουμε, να διαδώσουμε σωστά και να δημοσιοποιήσουμε στο κοινό, στις χώρες ειδικά αυτές, τις επιτυχίες αλλά και σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καμιά φορά εμπνέομαστε κι εμεί για να έχουμε τις αντίστοιχε μεταρρυθμίσει Σε έναν ε, παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ε, η αυξημένη ανταγωνιστικότητα, ε, οι δημόσιες πολιτικές, η διοίκηση, τα θέματα εξωτερικής ασφάλειας και, και εξωτερικής πολιτικής είναι ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Συνολικά, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι σε συνεργασία με τους Σκιώδης που ήδη συνεργάζονται μαζί μου σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, θα έχουμε μια ουσιώδη συμβολή με τις τροπολογίες που θα κατατεθούν Βέβαια, υπάρχει μία μη ρεαλιστική προθεσμία, 26 Φεβρουαρίου. Να προτείνω να πάει η προθεσμία την Τρίτη, μετά την Πράσινη Εβδομάδα, για να μπορέσουμε η δουλειά που θα κάνουμε να είναι πιο σωστή και όχι τόσο αγχωτική. Καλό λοιπόν τα μέλη της ΑΦΕΤ να μου καταθέσουν τα σχόλιά τους, ειδικά τους σκιώδης που βλέπω εδώ στην αίθουσα ε, και θα τα ακούσουμε με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ για την επέκταση της προθεσμίας να ελέγξουμε. Ίσως να μην υπάρχει αρκετός χρόνος πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Να το, το ελέγξουμε λίγο, να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ για την σύσταση, τις ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις. Τώρα έχουμε τους σκιώδεις. Ο κύριος Σικόφσκι είναι ο στην λίστα μου, εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την πολύ καλή σύνοψη, ικανότατη σύνοψη. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι η ανατολική εταιρική σχέση ε, είναι μια επιτυχία, είναι ας πούμε το κληροδότημα της Πολωνίας και της Προεδρίας της, ένα πρόγραμμα που πρότεινε Πολωνία και Σουηδία και που επηρέασε τη ζωή των ανατολικών εταίρων μας. Ε, δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν στην διαχείριση των συνόρων, σε πρωτοβουλίες ε, για διασυνοριακό τουρισμό, ε, επιχειρήσει μέσα στα πλαίσια του Erasmus Plus και πάνω απ' όλα οι χώρες αυτές έχουν αλλάξει τα εσωτερικά τους ε, σε τέτοιο βαθμό που τελικά τρεις από αυτές πήραν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεώρηση. Και από ό,τι ακούω, Κατομμύρια πολίτες αυτών των χωρών έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα και έχουν τιμήσει τους όρους αυτής της πρόσβασης χωρίς βίζα με, εξωτε... με εξαιρετική ε, ικανότητα, με καλά αποτελέσματα. Δείχνουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν λοιπόν τους κανόνες. Να επικεντρωθώ στο more and more ε, και όχι στο less for less. Υπάρχει αυτή η αυτοδιαφοροποίηση μεταξύ των έξι, γιατί κάποιοι θέλουν να γίνουν μέλη και άλλοι όχι. Ξέρουμε τις πολιτικές πραγματικότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανατολική εταιρική σχέση δεν μπορεί να τους δώσει την ιδιότητα του μέλους, αλλά μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν υποψήφιες χώρες, ε, βοηθώντας να εξυγχρονιστούν. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι θα πρέπει να ψάξουμε και άλλους τρόπους για να συνεργαστούμε με τους έξι. Πέρα από τον, ε, σφαίρα της ενέργειας που αναφέρατε ότι είναι κρίσιμη, το επόμενο μεγάλο project ε, θα πρέπει να είναι τα δεδομένα. Και ο κανονισμός για την ιδιωτικότητα των δεδομένων Ο υπερχόμενος κανονισμός για τον κυβερνοχώρο ε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά. Ελπίζω λοιπόν, χαίρομαι για την πρόοδο και ελπίζω ότι τα μέλη της ανατολικής εταιρικής σχέσης δεν θα έχουν σε αυτή τη σχέση την τελευταία μορφή σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κύριος Αντορόια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, συναδελφοί. Δυστυχώς ο, ε, ο εισηγητής, ο κύριος Σκόβατς, δεν βρίσκεται εδώ. Γι' αυτό θα τον αντικαταστήσω και να παρουσιάσω τη θέση μας. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα πολύ περιεκτικό κείμενο. Συμφωνούμε πάρα πολύ ε, και ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή που ετοίμασε αυτό το πολύ περίπλοκο και συνολικό κείμενο. Συμφωνούμε ότι η εταιρική σχέση είναι πολύ σημαντική από την άποψη της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άποψη της ασφάλειας και της οικονομίας των χωρών της εταιρικής σχέσης. Ε, η εκθεσή ε, ε, αναγνωρίζει τις προσπάθειες των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής ε, Χώρας. Επίσης, εκτιμούμε ότι η έκθεση σύνστα βαθύτερη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ανατολική Εταιρικής ε, Σχέσης και, και ανάμεσα σε αυτές επίσης. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα όπως είναι η ε, καταπολέμηση της διαφθοράς, η κλιματική αλλαγή, η οικονομική ανάπτυξη, η ισότητα των φύλων, η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας επίσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό για την ομάδα των σοσιαλιστών να συμπεριλάβουν κάποια επιπρόσθετα σημεία στην έκθεση αυτή. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε ε, με την ευκαιρία ε, να, ε, να ενθαρρύνουμε την ευθυγράμμιση με τα άρθρα 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ένα από τα σημαντικότερα είναι η τήρηση του κράτους δικαίου. Με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι για την ε, διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες και τέλος αλλά όχι έσκατον θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι η ανατολική εταιρική σχέση δεν μπορεί να ε, είναι θέμα ε, του, διαλόγου που ε, είναι ριζωμένος στη διαφορετικότητα των χωρών μελών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλά προετοιμασμένη έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η σχέδιση συγγήτρια από πλευρά των Πρασίνων είναι η κυρία Μαρκέτα ε, Γκρεγκόροβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο σύσταση προ το Ευρωκοινοβούλιο. Η ενατολική εταιρική σχέση είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μετά την αναθεώρηση των 10 ε, χρόνων υπάρχουν αλλαγές που θα πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε μια ολιστική προσέγγιση προς τις χώρες αυτές, διατηρώντας ε, μια πόρτα ανοιχτή και στήριξη προς όλους τους εταίρους και όλες τις ενισχυμένες προοπτικές και τις εξατομικευμένες λύσεις. Ε, εξατομικευμένη προσέγγιση δεν σημαίνει ε, σχέση δύο ταχυτήτων, διότι το να αφήνουμε ε, κάποιες χώρες να μένουν πίσω ε, ε, φέρνουμε άλλε χώρες. Θα πρέπει να τονίσω ότι η μακροοικονομική ε, βοήθεια είναι επίσης σημαντική. Η βοήθεια που λαμβάνεται από την ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την εκδημοκρατοποίηση και τους θεσμούς για να στεθεροποιηθεί η γειτονία, τηρώντας επίσης τις αξίες και τους κανόνες. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε επίσης μια ε, στατηγική μακροπρόθεσμη δέσμευση ε, ε, επικεντρωνόμενη στην δημοκρατοποίηση. Η έλλειψη ε, δημοκρατίας ε, θα δημιουργήσει ανοιχτό χώρο για άλλους ανοιχτούς παίκτες. Θα πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία με άλλους συντελεστές, ε, με τις ίδιες ιδεολογίες, έτσι ώστε να μετριάσουμε τις αρνητικές επιδράσεις στην ανατολική γειτονία και να αντανακλούμε την παγκόσμια τάση ε, της προπαγάνδας που ε, αποτελεί ε, την δυσφήμιση και την παραπληροφόρηση. Εδώ αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα αυτών από την Ανατολική Εταιρική Σχέση να λάβουν μεταρρυθμίσεις και να ανταποκριθούν στα κριτήρια μας που μια μέρα θα είναι επιλέξιμα μέλη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει πλήρη υλοποίηση των τρεχουσών συμφωνιών ανάμεσα στι δύο πλευρέ. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι προσβλέπω στη συνεργασία με τον Σιγητή και τους άλλους σκιώδη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η σκιώδη ε, ε, εισηγήτρια για την Ισιάρη είναι η κυρία Άννα Φωτίγκα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, επί επιτρέψτε μου να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή μας, τον Πέτρας Αουστρεβίτσιους, για το περιεκτικό έργο που έχει επιτελέσει. Θα επαναλάβω αυτά που είπαν και οι προλαλήσαντες, εξολογώντας ε, το σχέδιο αυτό και τις επιτυχίες του σχεδίου και την αναγκαιότητα να ε, το ενισχύσουμε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ στο δικό μου τομέα ενδιαφέροντος, την ασφάλεια, τη γενική ασφάλεια και την άμυνα. Όταν α, ε, σκεφτόμαστε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια ή την ε, Σφαιρική Στρατηγική του 2016, ε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική όταν αναφερόμαστε στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, της, εταιρικής, της ανατολικής μας γειτονίας, που για πολλά χρόνια αντιμετωπίζουν ε, ε, την επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Χώρες όπως είναι η Ουκρανία που θα πρέπει να συνδυάσουν σκληρές μεταρρυθμίσεις ε, για αυτές η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ο ρόλος μας εδώ είναι να δώσουμε μια όθηση σε αυτές τις χώρες ε, για το όφελος του κρανικού λαού να ε, ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων. Μερικές φορές ίσως να φαίνεται σκληρό, αλλά είναι εξαιρετικά απαραίτητο για εκείνους ε, για να πετύχουν μια πραγματική συνοχή και να πλησιάσουν το επίπεδο ανάπτυξης των δικών μας κρατών μελών. Όταν αναφερόμαστε στη Γεωργία, η Γεωργία είναι μια μικρή χώρα που αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πολύ έντονη πολιτική κατάσταση. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη χώρα και τον λαό της Γεωργίας. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η κατάσταση εκεί. Γνωρίζω ότι η κοινωνία της Γεωργίας είναι ίσως η πιο φιλοδυτική σε όλο τον κόσμο. Ενώ ταυτόχρονα η κατάσταση εκεί είναι τόσο δύσκολη. Και θα πρέπει να συμβάλλουμε και ε, στις δύο χώρες και οι δύο χώρες συμβάλλουν στην κοινή ε, ασφάλειά μας. Έχουμε συμφωνίες σύνδεσης ε, με συμφωνίες πλαισίου που θεσπίζουν τη συμμετοχή τους στην ΚΕΠΑ και αυτό αναφέρεται επίσης και στη Μολδαβία. Ακόμη και αν υπάρχουν πολιτικές αλλαγές σε όλες τις χώρες, αυτή η συνεισφορά στην παγκόσμια ασφάλεια, στην κοινή ασφάλειά μας, είναι τεράστια και θα πρέπει να την επικροτήσουμε. Γνωρίζουμε το επίπεδο που ασκείται στη Λευκορωσία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ε, την περίπτωση της Λευκορωσίας και να στηρίξουμε την κοινωνία της Λευκορωσίας χωρίς κανένα δισταγμό και επιφύλαξη, όπου υπάρχουν πολλοί, πολλές δυσκολίες και περιορισμοί. Ε, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες εδώ, για την Αρμενία, για το Αζερβαϊτζάν, που επίσης ε, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και προσπαθούν να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να υπερπηδήσουν τους περιορισμούς που υφίστανται. Ευχαριστώ. Uh, <clears throat> Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, λοιπόν, έχω κάποιους ομιλητές. Ε, πρώτα απ' όλα η κυρία κυρία Κανιέτε, ναι, συγχαρώ τον κύριο Στραβίτσιους ε, στην πληρέστατη προσέγγιση του. Ε, στην ουσία έχει καλύψει όλες τις πτυχές, όλες τις συνιστώσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που είπαν ήδη οι συνάδελφοι, αλλά ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Γεωργία ε, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν διάφορες κατηγορίες. Ο πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός εξέτησε την ποινή του και είναι πλέον ελεύθερος και εμείς παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά ώστε να μην υπάρξει άλλη επανάληψη του φαινομένου Ουμπουλάβα. Τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή την πορεία της δημοκρατίας των χωρών της Ανατολικής Εταιρική Σχέσης. Ανησυχώ και για τη Μολδαβία και ανησυχώ ότι υποχωρεί η δημοκρατία στην Γεωργία. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την ερεσιμότητα όταν ενισχύουμε χρηματοδοτικά τις χώρες αυτές, όχι μόνο επί τη βάση τεχνικών προϋποθέσεων και κριτηρίων, αλλά και επί τη βάση της πολιτικής τους αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και την ικανότητά τους και βούλησή τους να υλοποιούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί ανησυχώ τόσο διότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση τους θέλουμε σταθερούς δημοκρατικούς γείτονες και συνεργάτες. Γιατί βλέπουμε ότι ε, εκλογή προς εκλογή υπάρχει μία ολίσθηση από και προς ε, ένα σταθερό δημοκρατικό καθεστώς ή λιγότερο δημοκρατικό. Πριν από λίγα χρόνια χρησιμοποιούσαμε πολύ συχνά έναν όρο, τώρα τον ξεχάσαμε κάπως. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρεί σχέσεις με τις ε, χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και πρέπει να είναι και σκληρή αλλά και στοργική, τα φλόβια να το πούμε ελληνικά. Γιατί όλα αυτά είναι υποφελή και για τη Γεωργία και για τη Μολδαβία και για άλλες χώρες στα Ανατολικά και πλησιάζοντας προς τη Σύνοδο εκφράζω την ελπίδα ότι αυτή η έκθεση μπορεί να συνεισφέρει και η Σύνοδος να δημιουργήσει ένα νέο όραμα για την όλη πολιτική της Ανατολικής Γειτονίας και Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Κουμπίλιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι τη της Euronest και έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη να βλέπουμε θέματα μεταξύ άλλων ανατολικής εταιρικής σχέσης όσο ενδελεχέστερα μπορούμε. Στα πλαίσια αυτής της ενδελεχούς εξέτασης χαιρετίζω την ε, έκθεση αυτή και συγχαίρω το συνάδελφο Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι τι θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε ενδεχομένως περισσότερο. Νομίζω ότι οι επόμενες φάσεις θα εξαρτηθούν πάρα πολύ σε μια ισορροπία αλλά και συμπεριληπτικότητα στη διαμόρφωση της πολιτικής της ανατολικής εταιρικής σχέσης. οι ανατολικές χώρες θα πρέπει να μετατραπούν σε ή μάλλον προκειμένου να μετατραπούν σε success stories θα χρειαστεί εμείς να προσφέρουμε κίνητρα καρότα λέει ο μιλητής προς τους λαούς, τους πολίτες αυτών των χωρών υποαιρέσεις Γιατί αν δεν μπορέσουμε να τους ε, δείξουμε ρεαλιστικά μία προσδοκία, μία πορεία ενταξιακή, θα πρέπει κάτι να τους δείξουμε. Και λέω να τους δείξουμε καρότα, αλλά με κριτήρια. Είναι σημαντικό να ακούμε τους ανατολικούς μας εταίρους και η Euronest είναι ακριβώς αυτό το χώρος που έχουμε δημιουργήσει ώστε να τους ακούμε. Ήθελα να θυμίσω ότι τρεις συνδεδεμένες χώρες με συμφωνίες δηλαδή σύνδεσης και ελευθέρων συναλλαγών, έχουν σημειώσει πρόοδο και θέλουν να δουν αυτή την αρχή του πιο πολύ για πιο πολύ στην πράξη. Στις 5 Δεκεμβρίου υπεγράφει μια επιστολή από τον υπέξ της Γεωργίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας όπου υπογραμμίζουν τις αρχές της διαφοροποίησης και καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συστήσει τον διάλογο με τις συνδεδεμένες χώρες. Ένα διαρθρωμένο δηλαδή διάλογο με τις συνδεδεμένες χώρες. Το more for θα πρέπει να γίνει πιο απτό και να δίδει κίνητρα για μεταρρυθμίσει σε, σε τέτοιες χώρες όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία. Γνωρίζουμε το πλαίσιο εντός του οποίου συμβαίνουν όλα αυτά, λέει ο αλλά και εμείς από πλευράς μας πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, δείχνοντάς τους τι θα μπορούσαν να χάσουν αν δεν συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν και άλλες χώρες, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές αυτές ανατολικής Τερικής σχέσεις, Ξέρουμε ότι η Αρμενία θέλει να προλάβει με αυτές τις τρεις, να προλάβει αυτές τις τρεις πιο προχωρημένες χώρες. Και αυτή η, αν θέλετε, το πιο υψηλό επίπεδο εταιρική σχέση θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό το καρότο που έλεγα. Επομένως εγώ χαιρετίζω την έκθεση αλλά θα ήθελα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ομάδες υποστήριξης για Γεωργία και Μολδαβία τι είδους. Επίσης θα ήταν καλό να εξετάσουμε πιο προσεκτικά όταν μιλάμε για την επόμενη δεκαετία την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, λέει ο για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξή τους. δηλαδή μέσα όπως χρησιμοποίησαμε και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Διασυνδεσιμότητα, πλατφόρμες επενδύσεων και τα λοιπά. Αυτή τη γλώσσα θα μου άρεσε να την δω και σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Κομπίλιος, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπασέσκου έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εδώ έχουμε μια εξαιρετική έκθεση. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω στην έκθεση, αλλά θα προσπαθήσω να συνεισφέρω καμιά καλή ιδέα. Πρέπει να επαναβεβαιώνουμε την δέσμευσή μας για την ολοκλήρωση της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να την ολοκληρώνουμε ποικιλοτρόπως. να κινήσουμε ένα πολιτικό όραμα, λέει ο μιλτής. με κίνητρα. Κίνητρο για αυτούς είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων, για παράδειγμα. Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί, να σκεπτόμαστε και το επόμενο βήμα. Γιατί αν η πρόοδος τους συνδέεται με νέα υποστήριξη, αυτό λειτουργεί. Αν δείτε τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Γεωργία, όλες αυτές οι χώρες έχουν κομμάτι του εδάφους τους που κατέχεται από τη Ρωσία, λέει ο υβριδικούς πολέμους που έχουν ξεκινήσει οι Ρώσοι. Γιατί να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί μας για την καταπολέμηση των απειλών αυτών, των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τα λοιπά. Σε τέτοια πράγματα πρέπει να συνεργαστούμε. Και για το συντονισμό των ε, χρηματοοικονομικών μέσων που έχουμε, πρέπει να εστιαστούμε σε ουσιαστικά έργα υποδομών, ενέργειας μεταφορών, της ψηφιακής τεχνολογίας για να πλησιάζουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Υπάρχει η λέξη ντοντών που εκφράζει το φιλορωσικό πολιτικό ρεύμα στη Μολδαβία το οποίο όμως δεν κάνει κάτι για να εναντιωθεί σε αυτά τα βήματα του πλαισίου της ε, εταιρικής σχέσης. Δηλαδή ακόμα και ένας φιλορώσος ηγέτης μπορεί να προχωρήσει προς μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μου λένε ότι ο κύριος Λόρις Μέντιθ εκπροσωπεί εδώ την ε, γάμα δέλτα Νίερ. Θα θέλατε το λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματικά χαρά μου που βρίσκομαι ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της Ανατολικής Γειτονίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αουστρεβίτσιους για την ξεκάθαρη έκθεσή του. Επιβεβαιώνω ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής σε συνεργασία με την ΕΙΑΣ είναι προτεραιότητα όλα αυτά ε, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου. Θα είμαι σύντομος γιατί τα περισσότερα έχουν υποθεί. Είχαμε διαβουλεύσεις μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, χάρη στο Κοινοβούλιο και τις πληροφορίες του που μας έδωσε είχαμε πάνω από 200 συνεισφορές από κράτη-μέλη, χώρες στη εταιρική σχέση. Ε, υπήρξαν λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις ε, στον είπα αρμοστή και στην Κομισιόν ε, που θα κατατεθούν στα τέλη του Μαρτίου ως βάση για τις συζητήσεις που θα γίνουν στη Σύνοδο Κορυφής. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, φαίνεται ότι η κατεύθυνση ε, που πήραμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 ήταν η σωστή. Περισσότερη διαφοροποίηση. Ευχαριστούμε. Μεγαλύτερη ιδιοκτησία. Εργαζόμαστε από αυτού. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, αλλά γενικά ε, με το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη δίνουμε έμφαση σε αυτό επικεντρωνόμαστε σε μια ξεκάθαρη ημερήσια διάταξη που συμφωνήσαμε ε, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης 20 παραδοθέντα για το 2020 και επίσης η δημιουργία της ε, ε, ομάδας υποστήριξης για την Ουκρανία, το Task Force, όλα αυτά σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μαζί με πυλώνες για την συνδεσιμότητα τους ανθρώπους, τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια. Γενικά υπάρχει το αίσθημα ότι η βάση αυτή είναι σταθερή, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Δίνεται περισσότερη έμφαση τώρα στο θέμα της ασφάλειας γιατί χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και τέλος υπάρχει η αίσθηση ότι χρειαζόμαστε ενισχυμένη προσέγγιση σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Ε, επίσης ε, για την νεολαία, το φύλλο, την ψηφιακή οικονομία. Η οικονομία και η συνδεσιμότητα νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Και συνολικά βλέπουμε μια αντίσταση, μια ανθεκτικότητα οικονομική, αλλά και σε δημοκρατικό θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο περιβαλλοντικό και σε επίπεδο κοινωνίας. Στι χώρες αυτές. Άρα, πολύ ισχυρή πρόταση, πολλές από τις ιδέες που με μεγάλη φράδια εξέθεσαν οι εισηγητέ έχουν μπει ε, σε αυτό το σχέδιο και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεισφορά σα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάρτα Βιτρικόφσκα, που είναι επικεφαλής της ομάδας για την Ανατολική Γειτονία, εκπροσωπεί την ΕΙΑΣ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να βρίσκομαι σήμερα εδώ στα πλαίσια της προετοιμασίας ε, της Συνόδου Κορυφής ε, και ε, του σχεδίου της σύστασης του Κοινοβουλίου για αυτή την Σύνοδο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο στη συζήτηση για το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ήδη πολλά έχουν υποθεί. Απλώς θα επαναλάβω αυτό που ο Λόρες Μέρντιθ ε, ήδη είπε. Η Σύνοδος Κορυφής θα λάβει χώρα στις 18 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Αναμένεται να εξεταστούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ε, σε σχέση με την τελευταία Σύνοδο Κορυφής το 2017 αλλά να δούμε και τη μεγαλύτερη δέσμευση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της, ε, αλλά και τις μελλοντικέ μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ε, της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Όπως υπόθηκε, πέρυσι υπήρξε μια διαρθρωμένη διαδικασία διαβούλευσης, ε, σκέψης δηλαδή, για την ανατολική εταιρική σχέση μετά το 2020 από τη δική μας πλευρά υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που βγαίνουν από αυτή τη διαδικασία και θα τα δείτε και στην κοινή ανακοίνωση για το μέλλον της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Αυτή τη στιγμή την ετοιμάζουμε και θα εγκριθεί τον επόμενο μήνα. Η ανατολική εταιρική σχέση έχει κάνει ε, πολλά πράγματα σε επίπεδο οικονομίας, σε επαφών μεταξύ ανθρώπων, ε, υπάρχει όθεση στον τομέα της διακυβέρνησης, του δικαίου, ε, πάταξη της διαφθοράς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικαιοσύνης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία, υπάρχει επιτυχία στους πυλώνες της συνεργασίας, υπήρξε ένας πιο επικεντρωμένος οδικός χάρτης με παραδοτέα για το 2020 με απτούς στόχους και αποτελέσματα που αναμένονται. Επίσης, εφόσον ε, παραμένει ε, σταθερή η αρχιτεκτονική, όλα αυτά σημειώνονται, σημειώνονται τα όσα είπατε και θα σκεφτούμε ε, να τα συμπεριλάβουμε στη μελλοντική ανακοίνωση για την ανατολική γειτονία, εταιρική σχέση, συγγνώμη, που θα εγκριθεί ε, τον Ιούνιο του, 2000, 2020. Ε, Ευχαριστούμε την κυρία Βιτρικόφσκα. Πάμε πάλι στον κύριο Πέτρα Σαουστρεβίτσιου, στο βασικό μας εισηγητή. Μπορείτε να σχολιάσετε τις ιδέες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους σκιώδη εισηγητές, για πολύ σχετικά σχόλια και εισηγήσει και αξιόλογα. Αυτό που αποκομίζω από τη σημερινή συζήτηση είναι ότι οι πολιτικές προϋποθέσεις θα θα πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιήσουμε, να μην το ξεχάσουμε ποτέ, διότι θέλουμε να έχουμε μια εταιρική σχέση ανάμεσα σε ίσους. Πώς μπορείς να έχεις αυτού του είδους εταιρική σχέση αν δεν ε, ε έχεις τις κυριότερες πολιτικές προϋποθέσεις εκεί. Δεύτερο, δεν πρέπει να περιοριστούμε ε, ε, σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, τα προγράμματα. Ε, πλατφόρμες συνεργασίας κλπ. Ένα πράγμα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι πολύ ειδικό για τις χώρες ε, της ανατολικής εταιρικής σχέσης, Γιατί ίσως να πρέπει να επεκτείνουμε υφιστάμενε γραμμές πολιτικής μέσα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλέσουμε αυτές τις χώρες να ενταχθούν και να γίνουν εταίροι στα εφιστάμενα. Για παράδειγμα, η Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal. Εγώ είμαι εναντίον στο να δημιουργήσουμε μια άλλη πράσινη πολιτική, μια πρόταση για τις χώρες της εταιρικής εταιρικής σχέσης. Έχουμε μια τόσο ολοκληρωμένη περιεκτική προσέγγιση στη ΕΕ, θα μπορούσαμε να τις καλέσουμε αυτές τις χώρες να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στην πολιτική της πράσινης ε, συμφωνίας, ε, λαμβάνοντα υπόψη τις οικονομικές τους δυνατότητες και την πρόοδο. Αλλά ας μην δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό και ειδικό. Δεν είναι ειδικέ περιπτώσεις είναι ισότιμες με εμά και είναι διατεθειμένες να συμβάλλουν όσο μπορούν. Και τέλος, Πρόεδρε, Νομίζω ότι ε, είμαστε στο είδο μήκο κύματος. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις μελλοντικές επιτυχίες της ε, ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης. Γι' αυτό ε, τίνουμε μια χειρά συνεργασίας και οι χώρες αυτές δεν είναι απλά γείτονες, είναι εταίροι μας. Εάν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, νομίζω θα πετύχουμε κάτι την επόμενη δεκαετία που ξεκίνησε ήδη από το 2009 επί Πολωνικής Προεδρίας με μια τόσο καλή πρόταση και ελπίζω μέχρι το 30 να, να είμαστε ακόμη ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματά μας και την ένταξη των χωρών της Ανατολικής Αττικής Σχέσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καταλακτικά σας σχόλια. Αναρωτιέμαι εάν το πακέτο της πράσινη Συμφωνίας θα μπορούσε να θεωρηθεί από αυτούς ως αμοιβή ή ως το καρότο όπως λέγαμε και πριν. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση προτάσεων. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 26 Φεβρουαρίου. Σημειώσαμε την ιδέα παράτασης αυτής της προθεσμίας. Θα δούμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και θα σας ενημερώσουμε στον έφτατο χρόνο. Ας κλείσουμε και αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο είναι τα διάφορα. Δεν βλέπω οποιαδήποτε διάφορα και το τελευταίο μας σημείο είναι η προσεχή συνεδριάσεις. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής είναι η 16 Μαρτίου εδώ στις Βρυξέλλες και η 17η Μαρτίου επίσης εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σύνοδο. Ε, κυρίσω τη λήξη της συνόδου.